Bueno, Λοιπόν, μέχρι να φτάσουν οι συνάδελφοι, θα δούμε ένα βίντεο που θέλω να το δείτε πριν αρχίσει η συνεδρίαση.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 τους άλλους εκπροσώπους που είναι εδώ στο Προεδρείο και θα τους ε, παρουσιάσω όπως θα παίρνουν το λόγο τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εργασία που επιτελούν. Έχουμε εδώ τον κύριο Πλέκοβιτς που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και να του δώσω το λόγο για να κάνει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί ε, συνάδελφοι, ε, αγαπητές κυρίες, προσκεκλημένοι της ε, σημερινής ακρόασης και υπεύθυνοι της εκστρατείας για τα ε, παιδιά. Θα ήθελα να σας χαιρετήσω εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, εκ μέρους του κυρίου Μπρόκ συγκεκριμένα, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας σήμερα, οπότε μου ζήτησε να σας μεταφέρω το χαιρετισμό του και την εκτίμησή του για τη δουλειά σας στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ε, τα δύο βασικά νούμερα ε, που αφορούν ε, ε, τα παιδιά τα τελευταία δέκα χρόνια, δύο εκατομμύρια παιδιά περίπου έχασαν τη ζωή τους σε ένοπλες συγκρούσεις. Σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον 300.000 παιδιά στρατιώτες σε όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά σοκαριστικά αυτά τα νούμερα και θα έπρεπε να μας ανησυχούν πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι η προώθηση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών είναι προτεραιότητα της ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της κοινή εξωτερικής πολιτικής, αναπτυξιακής ε, πολιτικής, όπως επίσης και της ανθρωπιστικής ε, βοήθειας. Τα εργαλεία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολλαπλά και αλληλοσυμπληρούνται. Υπάρχει ο πολιτικός διάλογος, η πολυμερή συνεργασία, οι επιχειρήσει διαχείρισης ε, κρίσεων, ε, ε, η ειδική κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. Θα ήθελα ε, να ε, δείξω σήμερα στους προσκεκλημένους μας σε ποιο βαθμό ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ συνεργάζονται για το θέμα αυτό, πόσο αποτελεσματική και πόσο βαθιά είναι η συμπληρωματικότητα μεταξύ των εργαλείων και των οικονομικών μέσων που έχουμε για να αναλάβουμε τις δραστηριότητές μας. Ποιες θα μπορούσε να είναι, πόσο, πόσο περισσότερη θα μπορούσε να είναι η σύνδεση των προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των, του παιδιών στρατιωτών ε, και τα δεδομένα τα οποία ανέφερα προηγουμένως ε, μαζί με το ε, εντυπωσιακό βίντεο το οποίο ήταν πραγματικά επί της ουσίας και είναι κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα σε πολλά μέρη του κόσμου. Η, εκμετάλλευση των παιδιών σε πάρα πολλών παιδιών σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, επηρεάζει τις ζωές και των παιδιών αλλά και ε, γυναικών και ανδρών, παιδιών που δεν ζουν τη ζωή τους όπως εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τέλος πάντων στο ε, δυτικό ε, κόσμο θα θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να τη ζουν. Ε, χαιρετίζω λοιπόν την πρωτοβουλία της κυρίας Βαλενθιάνο ε, ως Προέδρου, ε, όπως επίσης και όλων των προσκεκλημένων για τις προσπάθειές τους ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Εκφράζουμε λοιπόν την εκτίμησή μας εκ μέρους ολόκληρης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λέλα Ζερβούγκη που είναι ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για τα παιδιά τα οποία θίγονται από ένοπλε συγκρούσει. Κυρία Πρόεδρε τη Επιτροπή Ανθεκιβίων Δικαιωμάτων, και Πρόεδρε τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κύριοι προσκεκλημένοι, Επιτρέψτε μου καταρχάς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την οργάνωση της συνάντησης αυτής για την εξτρατεία παιδιά και όχι στρατιώτες που προσπαθεί να βάλει ένα τέλος στη χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών από τις κυβερνητικές δυνάμεις που βρίσκονται σε ένοπλες συγκρούσεις. με στόχο να προστατευτούν τα παιδιά από αυτές τις συγκρούσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη για την διαρκή τους υποστήριξη προς το πρόσωπρό μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη ποτέ δεν παρέλειψαν να υποστηρίξουν δημοσίως τα παιδιά και τι τις προσπάθειες που καταβάλει η κοινωνία των πολιτών και το Ηνωμένα έθνη για να προστατεύσουν τα παιδιά που έχουν βρεθεί στα γρανάζια των ένοπλων συγκρούσεων. Κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους πολλά παιδιά και πολλές οικογένειες σαν αποτέλεσμα συγκρούσεων. Τα παιδιά, όλα αυτά έχουν κάτι κοινό. Περνάνε χρόνια ολόκληρη τη ζωή τους ενδεχομένω προσπαθώντας να συνέλθουν από την κακοποίηση αυτή. Τα τραύματά τους είναι ψυχολογικά και σωματικά. Η θέση μου δημιουργήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μετά από την ε, δημοσίευση το 1976 της έκθεσης σχετικά με την επίπτωση που έχουν οι ένοπλες συγκρούσεις στα παιδιά. Η έκθεση αυτή απεκάλυψε στον κόσμο το εύρος της χρήσης των παιδιών στρατιωτών και τη σοβαρότητα που έχει κάτι τέτοιο. Έδειξε την σε ανάλογη επίπτωση που έχουν οι ένοπλες σειράξεις στα παιδιά και θεώρησε ότι είναι τα βασικά θύματα των ένοπλων συγκρούσεων. Η έκθεση αυτή έγινε δεκτή από τη διεθνή κοινότητα ως μία έκκληση για δράση και για ενδυνάμωση των μηχανισμών προστασίας των παιδιών. Από το 1999 υπάρχει συστηματική δέσμευση του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο ε, έθεσε την προστασία των παιδιών που θίγονται από τις ένοπλες συγκρούσεις στην καρδιά της ημερησίας διάταξη ε, για θέματα ειρήνης και ασφάλειας διεθνούς χαρακτήρα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, μας έδωσε ένα νομικό στέρεο πλαίσιο καθώς και τα εργαλεία για να τεκμηριώσουμε, να καταγγείλουμε και να απαντήσουμε στις ε, παραβιάσεις που αφορούν τα παιδιά. Καταρχάς το Συμβούλιο όρισε έξι σοβαρά δικήματα που επηρεάζουν τα παιδιά σε περίοδους σύγκρουσης. Την ε, χρήση των παιδιών την ε, ε, τον ακροτηριασμό και τη δολοφονία παιδιών, τη σεξουαλική βία που ασκείται κατά των παιδιών, ε, επιθέσεις ε, κατά των σχολείων και των νοσοκομείων, την παρεμπόδιση ανθρωπιστικής βοήθειας και την σύλληψη παιδιών. Το Συμβούλιο υιοθέτησε ψηφίσματα βάσει των οποίων ζητούντο τα παρακάτω στα Ηνωμένα Έθνη. Πρώτον, να συγκεντρωθούν και να επιτευχθούν πληροφορίες, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς τα παιδιά επηρεάζονται από τις ένοπλες συγκρούσεις και να χρησιμοποιηθούν αυτές οι ε, πληροφορίες για να προετοιμαστεί και να υποβληθεί μια ετήσια έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Συμβούλιο επίσης ζήτησε να, να εντοπιστούν και να ε, τα μέρη της σύραξης ε, τα οποία χρησιμοποιούν ε, τα παιδιά και τα σκοτώνουν και τα ε, ακροτηριάζουν. Τέλος, μας ζήτησε να ξεκινήσει ένας επικοδομητικός διάλογος με τις κυβερνήσεις καθώς και με τις ένοπλες ομάδες που είναι καταγεγραμμένες έτσι ώστε να υπάρξει ένα πρόγραμμα δράσης για να τεθεί τέλος και να προληφθούν οι παράνομες αυτές δράσεις κατά των παιδιών. Τα προγράμματα δράσης συμπεριλαμβάνουν μια σειρά από απτά μέτρα για τις καταγεγραμμένες ομάδες, είτε είναι κρατικές είτε δεν είναι κρατικές, με στόχο να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά. Συγκεκριμένα απτά μέτρα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να σταματήσει η βία κατά των παιδιών για να μπορέσουν να απελευθερωθούν και για να μπορέσει να εξασφαλιστεί μια μακρά διάρκεια επανένταξή τους αλλά και για να δημιουργηθούν μηχανισμοί για να προληφθεί η ε, χρησιμοποίηση των παιδιών για, ε, σε ένοπλες συγκρούσεις καθώς και η στρατολόγησή τους. Για, την, ε, για να μπορέσει να σε εφαρμογή ε, τη εντολή, το γραφείο μου εργάζεται στενά με το σύνολο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης και της UNICEF, αλλά η ΕΤΕ, έχουμε και εταίρους στην κοινωνία των πολιτών, περιφερειακές οργανώσεις και υποπεριφερειακές οργανώσεις, όπως α πούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ανοίγει στι περιφερειακές οργανώσεις, ενώ υπάρχει η ενεργό στήριξη πολλών χωρών. Ορισμένες χώρες ε, έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή από τις άλλες, όπως σας είπα, ένα σημαντικός μας εταίρος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί τόπου εφαρμόζονται προγράμματα δράσης και συντονίζονται από μια ειδική ομάδα κρούσης όπου συμπροεδρεύει η ύπατη ε, αρχή που εκπροσωπεί τα Ενωμένα Έθνη στη χώρα και ένας εκπρόσωπος της UNICEF. Έχουμε στην ημερησία μας διάταξη 23 περιπτώσεις ένοπλων συγκρούσεων που είναι εγγεγραμμένες στο χρονοδιάγραμμα των, του Γενικού Γραμματέα και που αφορούν παιδιά που εμπλέκονται σε συγκρούσεις. Έχουμε 59 περιπτώσεις περιπτώσεις οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τα δικήματα που σας παρέθεσα. Εκτό από αυτές είναι δυνάμεις και κυβερνητικές δυνάμεις, ενώ 50 ε, μία είναι μη κρατικέ οργανώσεις. Μεταξύ των 23 αυτών περιπτώσεων θα πρέπει να συγκρίνουμε έξι περιπτώσεις μίζωνος κρίσης, όπου συμπεριλαμβάνονται ομάδες όπως η Άιζιλ και την Μπόκο Χάραμα, που γνωρίζετε τι συμβαίνει με τα παιδιά. Και αυτό είναι μόνο μία περίπτωση των όσων υφίστανται. Οι ομάδες αυτές χρησιμοποιούν τακτικές ακραίας βίας και πάρα πολύ συχνά τα παιδιά αποτελούν έμεσα ή άμεσα θύματα. Όπως αναφέρθηκε ήδη εδώ και μερικές μέρες γιορτάσαμε την 25η επέτειο από την ε, ε, υιοθέτηση της Σύμβασης των ε, Δικαιωμάτων των Παιδιών. Είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε διανύσει μια μακρά πορεία για να βελτιωθεί η κατάσταση των παιδιών, κυρώνοντας τη Σύμβαση 184 αναγνωρίζουμε ότι τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια έχουν δικαιώματα και ότι οι κυβερνήσεις είναι οι υπεύθυνε για το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων αυτών. Παρόλα αυτά, η πρόοδος που κατεγράφει τα τελευταία 25 χρόνια είναι άνηση σε καιρό όλα τα παιδιά συνεχίζουν να δολοφονούνται, να κροτηριάζονται, να στρατολογούνται, να χρησιμοποιούνται από ε, ε, στρατηγικές δυνάμεις για να μην έχουν πρόσβαση στην υγεία και στην παιδεία. Παρόλες τις προσπάθειές μας, τα συμπεράσματα της ε, Γκράσα συνεχίζουν να είναι επίκαιρες. Στα ταξίδια μου στις ε, ζώνες συγκρούσεων συναντάω πολύ συχνά παιδιά που υποχρεώνται να καταλήψουν τα σπίτια τους μερικές φορές χωρίς τις οικογένειές τους. Πρόσφατα ε, στο Νότιο Σουδάν συνάντησα ένα μικρό αγοράκι που στην αρχή της πρώτης κρίσης στο Σουδάν βρέθηκε και σε λάθος μέρος τη λάθος χρονική στιγμή. Επτά μήνες αφού τραυματίστηκε είχε, ε, δυσκολευόταν να περπατήσει και ε, συνέχιζε να αγνοεί που βρίσκεται η οικογένειά του. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό για ένα παιδί. Παρ' όλα αυτά προσπάθησε να συνεχίσει τη ζωή του ε, σε ένα κέντρο για παιδιά του που ανήκει στα Ηνωμένα Έθνη. Ε, αποτελεί, ε, είναι ένας από τους τυχερούς που έχουν την ευκαιρία να ε, φιλοξενηθούν σε ένα τέτοιο κέντρο. Δεν συμβαίνει όμως αυτό πάντοτε. Κυρίες και κύριοι, παρόλες τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, η εμπλοκή μας σε αυτό το τομέα αρχίζει να αποφέρει καρπούς. Θα μπορούσαμε τώρα πλέον να πούμε και μπορώ να το πω έχοντας εργαστεί το, τόσα χρόνια ότι αρχίζει να διαφαίνεται μια συνένεση μεταξύ των κυβερνήσεων ότι και να συμφωνούν όλοι ότι τα παιδιά δεν έχουν καμία θέση σε ένοπλες συγκρούσεις. Σαν αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας ξεκίνησα την εκστρατεία «Παιδιά, όχι στρατιώτες» από κοινού με τη UNICEF για να μπορέσει να μπει τέλος η στρατολόγηση των παιδιών από τις ένοπλες κυβερνητικές δυνάμεις τη στιγμή που ξεκίνησε η εκστρατεία, οκτώ ε, ε, κυβερνητικά στρατεύματα είχαν καταγραφεί στα παραρτήματα της ετήσιας έκθεσης του Γενικού Γραμματέα για τα παιδιά ε, σε ένοπλες συγκρούσεις. Οι χώρες αυτές είναι το Αφγανιστάν, το Τσάντ, η, δημοκρατική, η Δημοκρατία του Κονγκό, το Μιανμάρ, η Σομαλία, το Σουδάν, ε, το Νότιο Σουδάν, το Σουδάν και η Εμένη. Οι κυβερνήσεις αυτές ήταν ε, μαζί μας τη στιγμή που ξεκίνησε η εκστρατεία για να μπορέσουν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος από αυτούς παρόν εδώ, αλλά θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να τους ευχαριστήσω. Επτά από αυτές τις χώρες προσυπέγραψαν προγράμματα δράση με, τις Ηνωμένες, ε, με τα Ηνωμένα Έθνη για να μπορέσει να μπει τέλος στην στρατολόγηση των παιδιών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι κυβερνήσει αυτές εξέφρασαν την επιθυμία τους να ακολουθήσουν μια διαφορετική πορεία σε ό,τι αφορά τη στρατολόγηση των παιδιών. Τα Ηνωμένα Έθνη ε, ε, έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να υποστηρίξουν Αυτέ αυτές τις προσπάθειες στην όλη διαδικασία εφαρμογή των προγραμμάτων δράση. Προσωπικά ε, συνεργάστηκα με τη UNICEF έτσι ώστε οι χώρες αυτές να έχουν πρόσβαση στους πόρους και την απαραίτητη τεχνική ε, ε, βοήθεια όχι μόνο για να προχωρήσει αλλά για να συμπληρωθεί, να περατωθεί αυτή η εφαρμογή των προγραμμάτων δράση. Γι' αυτό το λόγο η δική σας στήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εννέα μήνες μετά την έναρξη της εκστρατείας έχουν καταγραφεί σημαντικές πρόοδοι. Τον Μάιο η κυβέρνηση της Ιεμένης Φέτος το Μάιο υπέγραψε ένα πρόγραμμα δράσης με, τις με τα Ηνωμένα Έθνη. Με την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών το Τσάντ ολοκλήρωσε το πρόγραμμα δάσης και το εθνικό του στρατός απεσύρθη από τον κατάλογο του Γενικού Γραμματέα. Η κυβέρνηση του Αφγανιστάν υιοθέτησε ένα φύλλο πορείας για να επιταχυνθεί η εφαρμογή του προγράμματος ε, δράσης. Γιατί αυτός είναι ένας τρόπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για σας, τις χώρες μέλη, για να δείτε τι θα μπορούσατε να κάνετε σε αυτή τη χώρα. Το Μιαμάρα καταγράφει μια πρόοδο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος δράσης και απελευθέρωσε 373 παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Σομαλία δημιούργησε μηχανισμούς για να μπορέσουν να μεταφερθούν στα Ηνωμένα Έθνη παιδιά που ε, εντοπίστηκαν μέσα στα στρατεύματα και δημιούργησε μια ε, μονάδα προστασίας της παιδικής ηλικίας στις ένοπλες δυνάμεις. Η κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάνα αποφάσισε να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα δράσης. Φέτος, σε μια συνάντηση 29 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Άμυνας ανήγγειλε δημόσια ότι θα ελέγχεται η ηλικία των στρατιωτών σε όλα τα στρατόπεδα του SPLA που είναι ο στρατός του Νότιου Σούνταν στην ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό η κυβέρνηση διόρισε έναν προσωπικό εκπρόσωπο ε, του ε, Προέδρου του κράτους για να ενισχύσει την καταπολέμηση των σεξουαλικών βιοπραγιών και το, τη στρατολόγηση των παιδιών. Η κυβέρνηση μου ανακοίνωσε μια έκθεση αναλυτική των μέτρων που λήφθηκαν ε, από το 2013 όταν υπήρξε μια συμφωνία με τα Ηνωμένα Έθνη και υπάρχει αυτή η πρόοδος, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και, το Συμβούλιο Ασφαλείας στηρίζουν αυτήν την ε, εκστρατεία. Ο Αραβικός Σύνδεσμος, η Αφρικανική Ένωση και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στηρίξει τους στόχους. Και θέλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σε ευχαριστήσω για αυτή σας τη δέσμευση. Επίσης ενθαρρύνομαι από τις πρόοδους αυτές, από την υποστήριξη και τη δυναμική που δημιουργεί η εκστρατεία. Αλλά δύο χρόνια πριν από τη λήξη του προγράμματος ε, πολλά πρέπει ακόμη να κάνουμε για να είμαστε βέβαιοι ότι τα παιδιά προστατεύονται από τη στρατολόγηση στις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας των χωρών αυτών. Να μην ξεχνάμε ότι στις χώρες αυτές, σε αυτές τις 7 χώρες, Υπάρχουν επίσης 32 ένοπλες ομάδες οι οποίες στρατολογούν παιδιά. Άρα δεν είναι μόνο οι 7 κυβερνητικοί στρατοί. Αυτοί δημιούργησαν ένα πλαίσιο, αλλά πρέπει επίσης να μας απασχολήσουν και αυτές οι 32 ένοπλες ομάδες. Πρέπει να λήξει η βία στρατολόγηση των παιδιών από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Είναι δυνατόν κατά τα επόμενα δύο έτη, αλλά μόνο αν εργαστούμε από κοινού και μόνο εάν τις βοηθήσουμε μέσω της πείρας και των πόρων που μπορούμε να τους δώσουμε. Κύριοι βουλευτές, ε, διακεκριμένοι προσκεκλημένοι αγαπητοί συνάδελφοι, για να καταλάβετε καλύτερα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά σε συγκρούσεις και πώς μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο της εκστρατείας μας, θα, σας, ε, θα ήθελα να σας καλέσω να διατηρηθεί η ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πολιτική δέσμευση πρέπει να είναι εμφανής επιτόπου μέσω των πρεσβειών σας στις χώρες ε, όπου γίνεται αυτή η εκστρατεία αλλά και στις άλλες χώρες όπου τα παιδιά επηρεάζονται από ένοπλες συγκρούσεις. Πάντα επιτόπου στις χώρες αυτές η Ένωση θα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο στο συντονισμό και τη στήριξη στις ειδικέ ομάδες της κάθε χώρας που ε, εφαρμόζουν το πρόγραμμα δράσης για όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδιά που θίγονται από τι ανοπλέ συγκρούσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει να εγγυηθούμε μια βοήθεια στην πιο μακρά φάση, την πιο δαπανηρή φάση τη διαδικασία του προγράμματο δράση, Την επανένταξη των πρώην παιδιών στρατιωτών που πρέπει να γίνει με ψυχοκοινωνική βοήθεια, εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση για τους νέους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να μας δώσει την πείρα της, τη στήριξή της για να ενισχύσουμε την παροχή δικαιοσύνης, να ενισχύσουμε τις μεταρρυθμίσεις, να ενισχύσουμε την πάλη κατά της ασυδοσίας αυτών που βιοπραγούν κατά των παιδιών. Μόνο έτσι μπορούμε να προλάβουμε και να σταματήσουμε αυτές τις ε, βιοπραγίες και τις, ε, ε, τους βιασμούς. Ε, ξέρετε ότι το εφετείο του Διεθνούς Δικαστηρίου επιβεβαίωσε την απόφαση στην υπόθεση Λουμπάγκα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία. Επίσης πρέπει η προστασία των παιδιών να είναι ε, εγενές τμήμα των ε, συμφωνιών που κάνει με άλλες περιφερειακές οργανώσεις με την, Ευρωπαϊκή, με Αφρικανική Ένωση. Σε κάθε συνεργασία με την, Ευρωπαϊκή, με την Αφρικανική Ένωση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αυτή η συνεργασία και όπου είναι δυνατό η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει διαβήματα έναντι των κυβερνήσεων αλλά και έναντι άλλων εμπλεκομένων σε συγκρούσεις, ενόπλων ομάδων δηλαδή, για να σταματήσει αυτή η σοβαρή κακομεταχείριση. Η εκστρατεία «Παιδιά όχι στρατιώτες» μας δίνει τη δυνατότητα από κοινού να υλοποιήσουμε προγράμματα που θα έχουν πραγματική επίπτωση στη ζωή χιλιάδων παιδιών. Είμαι πεισμένη ότι είναι μια ευκαιρία που δεν θα αφήσουμε να μας ξεφύγει. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Σερούγκη. Τώρα να δώσουμε το λόγο, να δώσουμε το λόγο έλεγα, στην κυρία Γιώκα Μπραντ, που είναι η αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος των, των ΗΠΑ για τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχά, να συμφωνήσω με του προλαλήσαντε ε, που ευχαρίστησαν την Υποτροπή, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που οργάνωσε αυτή το ε, σημαντική συνεδρίαση σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκομαι εδώ σήμερα ε, με τους δύο ε, διακεκριμένους συναδέλφους με τους οποίους πραγματικά συνεργαζόμαστε πάρα πολύ επί θα ήθελα επίσης επί ε, τη ευκαιρία να αναφερθώ στο θέμα της στρατολόγηση των παιδιών ε, που πρέπει να το γνωρίσει καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι Ευρωβουλευτές σκεφτείτε να πηγαίνει κανείς ε, σχολείο, ε, λέει, γεια στους ε, φίλους του, αλλά δεν ξέρει ότι θα, γυρίσει, γιατί μπαίνει μέσα στην τάξη κάποιος, στην τάξη και απομακρύνει αυτό το παιδί από τους φίλους του. μετά τον ξυπνάνε τρεις ώρα το πρωί, ε, για να εκπαιδευτεί και τους δίνουν ε, να φάνε τρεις φορές την εβδομάδα. Φανταστείτε να, ε, να είναι κανείς τρομοκρατημένος και να έχει την επιλογή ή να καταδώσει και να σκοτώσει ή να καταδοθεί και να σκοτωθεί. Οπότε δεν μπορεί για σας να είναι πάρα πολύ περίεργο, αλλά ο Ντέιβιτ το έζησε αυτό. Ο Ντέιβιτ είναι 16 χρονών και ε, ζούσε ε, στο νότιο Σουδάν για τον Ντέιβιτ και για τις δεκάδες χιλιάδες ε, παιδιών στρατιωτών όπως εκείνος. Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από την 25η επέτειο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Είναι κάτι το οποίο ε, μας βρίσκει όλους υπεύθυνου. Πρέπει να είμαστε όλοι υπεύθυνοι και υπόλογοι για την ασφάλεια των παιδιών σε όλο τον κόσμο και εξασφαλίζει σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ε, θρησκευτικής ε, πεποίθησης, ε, ε, αναπηρίας, ε, φύλου, Εξασφαλίζει λοιπόν ε, ε, ασφάλεια, υγεία ε, για όλα τα παιδιά στον κόσμο. Πρέπει να γίνουν σοβαρές αλλαγές, όχι μόνο με ισχυρές δηλώσεις, αλλά και με ισχυρές πράξεις. Οπότε η UNICEF εκτιμά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σεβασμό όχι μόνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα, αλλά και των παιδιών και μέσω της εκστρατείας «Παιδιά, όχι στρατιώτες» συγκεκριμένα. Να ευχαριστήσω ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρόσφατο ψήφισμά του που τονίζει τη σημασία του να είναι ε, τα παιδιά το επίκεντρο της, ε, ε, του θεματολογίου μετά το 2015. Κάνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί ε, το θέμα ε, της αναπτυξιακής βοήθειας και το θέμα του δικαιωμάτων των παιδιών ε, πιο σφαιρικά. Γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία εξακολουθούν να στρατολογούνται και να χρησιμοποιούνται όχι μόνο ως στρατιώτες, αλλά ως κατάσκοποι, ως αγγελιαφόροι, ως μάγειρες. Πολλοί χρησιμοποιούνται ως σεξουαλικοί σκλάβοι ή κάνουν εξαναγκασμένους γάμους. Ε, πολλές φορές ε, ε, μέσω της, ε, και μέσω της UNICEF αλλά και μέσω άλλων ε, εταίρων μας μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Ε, ο Γενικός Γραμματέας χρησιμοποιεί μαρτυρίες στις εκθέσεις του στην, στο Συμβούλιο Ασφαλείας όταν ζητά από τις ενδιαφερόμενες χώρες να συμμορφωθούν με, τις, με τα διεθνή πρότυπα, με τις διεθνείς προδιαγραφές. Οι επτά κυβερνήσεις των χωρών εξακολουθούν να ε, μην ε, συμμορφώνονται ε, με, τις, με, τα αιτήματα της εκστρατείας παιδιά όχι στρατιώτες. Η κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το Νότιο Σουδάν και η Συρία είναι μεταξύ αυτών των χωρών. Πολλές φορές, για παράδειγμα, στις, Φιλικίνες, στις Φιλιππίνες το Ισλαμικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ε, δεσμεύτηκε να προστατεύσει τα παιδιά, αλλά αυτό που ισχύει για αυτούς δεν ισχύει υποχρεωτικά ούτε για του Εξέλεκα ούτε για τον Μποκοχαράμ. Οπότε ε, μερικές φορές ε, δεν υπάρχει πραγματική ε, βούληση συνεργασίας και όπως είδαμε υπάρχουν νέε νέες μορφές στρατολόγησης μέσω κοινωνικών ε, media μια στρατηγική βεβαίως την οποία εμείς καταδικάζουμε, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε νέους τρόπους ε, να ε, προλάβουμε αυτή την κατάσταση και νέους τρόπους να συνεργαστούμε. Παιδιά όπως ο Ντέιβιντ εξαρτώνται από το να κάνουμε εμείς ε, κάτι. Η η εκστρατεία αυτή πρέπει να επιτύχει και η UNICEF ε, θα κάνει ό,τι μπορεί για να ε, συμμετέχει ε, στο, επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσπαθούμε να επενδύσουμε σε προγράμματα υπέρ των κοριτσιών και των αγοριών για την προστασία και των παιδιών και για την καταπολέμηση Τη στρατολόγηση από ένοπλες ομάδε Θέλουμε να τα βοηθήσουμε να ε, ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Για παράδειγμα στο Αφγανιστάν, ε, στο, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στη Σομαλία, οι κυβερνητικές και οι τοπικές αρχές συνεργάζονται με τη UNICEF για να μπορέσουν 10-15 παιδιά να ξαναβρούν τι οικογένειε του και να επανενωθούν με αυτές. Ε, στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία επίση, ε, προσπαθούμε να ε, βοηθήσουμε τα παιδιά που έχασαν πάρα πολλά χρόνια από το σχολείο. Να μην ξεχνάμε ότι ενώ ε, ότι για τα παιδιά τα οποία βγαίνουν από αυτή την κατάσταση η εκπαίδευση δεν είναι μόνο ανάγνωση και γραφή, είναι ένας τρόπος να θεραπευθούν από τα τραύματά τους και να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας προσπαθούμε να προωθήσουμε ανθρώπους με δεξιότητες, ε, ε, ειδική κατάρτιση ή ε, μικρές επιχειρήσεις και να βοηθήσουμε ε, μέσω ε, συγκεκριμένων προγραμμάτων τα οποία δουλεύουν. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ε, περιοχών με ένοπλες συγκρούσεις. Όμως πρέπει να υπάρξουν διαδικασίες αξιολόγησης προκειμένου να μην υπάρξουν επιπλέον στρατολογήσεις. Πρέπει να υπάρχει καταχώρηση των παιδιών, ε, να, καταχωρούνται τα παιδιά, ε, τα διαβατήριά τους. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, γιατί ε, μπορεί η στρατιωτική βοήθεια να είναι πάντοτε υπό την αίρεση ε, της προόδου σε σχέση με τη μη στρατολόγηση παιδιών. Ε, και επίσης μέσω διάθεσης πόρων για την προστασία των παιδιών και ε, τη βελτίωση της ε, αποκατάστασης του. Ο Ντέιβιντ. ο David διέφυγε, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμη το ταξίδι του. Προσπαθεί ακόμη να βρει τροφή ε, και βασικά πράγματα όπως μία κουνουπιέρα και ένα σαπούνι. Θυμάται να παίζει ποδόσφαιρο, να πηγαίνει στο σχολείο και να βλέπει ταινίες. Ο Ντέιβιντ ε, δεν τα έχει παρατήσει, οπότε δεν πρέπει να τα παρατήσουμε κι εμείς. Ε, όσο αφιερωνόμαστε σε αυτή την προσπάθεια παιδιά, όχι στρατιώτες, ε, ας μας εμπνεύσει το κουράγιο του Ντέιβιντ και να πούμε ότι μια μέρα θα μπορέσουν παιδιά όπως ο Ντέιβιντ να βγουν από αυτή την κατάσταση και να έχουν ένα μέλλον ευημερία και ασφάλειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Lucy Withers που είναι σύμβουλος για ανθρωπιστικά θέματα της οργάνωσης Σώστε τα παιδιά, Save the Children. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να ευχαριστήσω την υποεπιτροπή για Ανθρώπινα Δικαιώματα του Κοινοβουλίου που μας κάλεσε, κάλεσε την οργάνωσή μας. Είναι τιμή που είμαστε μεταξύ των διακεκριμένων άλλων ομιλητών και ευχαριστούμε για την προσοχή της υποεπιτροπής σας και του Κοινοβουλίου γενικότερα για το θέμα των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις. Η προστασία των παιδιών από τα επιβλαβή αποτελέσματα των συγκρούσεων συμπεριλαμβανομένης ε, της στρατολόγησης και της χρήσης είναι βασικό στοιχείο της δουλειάς μας παγκοσμίω. Εργαζόμαστε συστηματικά σε χώρες όπως η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, η Κολομβία, η Μιανμάρ, το, το Νότιο Σουδάν ούτως ώστε να αποφευχθεί η στρατολόγηση και για να βοηθήσουμε την επανένταξη αγοριών και κοριτσιών που έχουν συμμετάσχει σε ενόπλες δυνάμεις, σε ενόπλες ομάδες. Δίνουμε βοήθεια για να υπάρχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και για να δοθούν ευκαιρίες. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τη διεθνή ανταπόκριση. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τη UNICEF με το γραφείο του ειδικού εκπροσώπου και γενικότερα με το σύστημα των ε, Ηνωμένων Εθνών για να προωθήσουμε διεθνείς προδιαγραφές, ε, βέλτιστες πρακτικές, όπου είναι δυνατό στην πράξη παρατηρούμε και κάνουμε εκθέσεις για σοβαρές παραβιάσεις συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, υποστηρίξουμε την ε, διατύπωση και εφαρμογή πολιτικών από περιφερειακά σώματα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνουμε και πολύ συγκεκριμένη βοήθεια, πρακτική βοήθεια. Για παράδειγμα σχεδιάζουμε και μεταδίδουμε έτοιμα προγράμματα για την επανένταξη σε διάφορες υπηρεσίες της Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, όπου υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις, τα παιδιά θα εμπλακούν. Είναι σχεδόν αναπόφευκτο. Όπως υπόθηκε, ο Γενικός Γραμματέας στην τελευταία έκθεση για το θέμα αυτό αναφέρεται σε 23 διαφορετικές καταστάσεις και αναφέρει 59 εμπλεκόμενους στις ένοπλες συγκρούσεις που ενεργά στρατολογούν και χρησιμοποιούν παιδιά σε ε, μάχες. Η χρήση των παιδιών έχει γίνει μόνιμη όπου ξαναρχίζουν οι συγκρούσεις, ξαναρχίζουν οι στρατολογίες παιδιών και η χρήση τους. Οπότε σήμερα ακόμη έχουμε μια κατάσταση όπου ανα πάσα στιγμή αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες παιδιών συμμετέχουν σε ένοπλες συγκρούσεις. Η κατάσταση αυτή δεν οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν αρκετές προδιαγραφές διεθνής νομοθεσία για το θέμα αυτό. Όπως είπε η ειδική εκπρόσωπος, υπάρχει σχεδόν παγκόσμια συνένεση ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς και έχουν επικυρωθεί οι διεθνείς συμβάσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα το θέμα αυτό και το θέμα αυτό απασχολεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, την Αφρικανική Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ενωμένα Έθνη. Όμως ε, η εφαρμογή δεν έχει προχωρήσει ακόμη και γι' αυτό το λόγο τα Ενωμένα Έθνη ξεκίνησαν αυτή την εκστρατεία που είναι τόσο σημαντική γιατί πρέπει να φωτίσουμε το θέμα αυτό και να στηρίξουμε τις δυνάμεις ασφαλείας των κρατών όπου υπάρχει λόγος για να εφαρμοστούν μέτρα για να σταματήσει η στρατολόγηση και να ε, επιστρέψουν ε, στην μη στρατιωτική ζωή τα παιδιά που είναι ήδη στρατολογημένα να απολυθούν από τις ενοπλές δυνάμεις. Πρώτα απ' όλα είναι περίπλοκο το θέμα της αντιμετώπισης της στρατολόγησης από μη εθνικούς στρατούς που είναι 51 από τις, ε, που είναι 51 από τις 59, 51 51 οργανώσεις που το κάνουν αυτό. Και θέλουμε επίσης σε μελλοντικές συγκρούσεις να μην υπάρχει στρατολόγηση ούτε από κυβερνητικού στρατού ούτε από άλλε ένοπλε ομάδε. Πρέπει με πολύ πιο ενεργό τρόπο να δούμε πού υπάρχει τέτοιο κίνδυνο και πιο αποτελεσματικά να τι αντιμετωπίσουμε. Όπω ήδη υπόθηκε, αυτό σημαίνει καλύτερη πρόληψη. Οι πολλοί, από του κίνδυνου είναι πολύ καλά κατανοητοί. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι οι νομικές απαγορεύσει στρατολόγηση και συμμετοχή των παιδιών δημιουργούν ένα ε, περιβάλλον θετικό, προστατευτικό Ξέρουμε ότι τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο όταν δεν μπορούν να αποδείξουν ε, την ηλικία τους, όταν η διαδικασία εξακρίβωσης ηλικίας στο σημείο στρατολόγησης είναι ανεπαρκής ή όταν ε, η πρακτική στρατολόγησης είναι άτυπη. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ποινικέ κυρώσεις ή η προσπάθεια είναι διαπιστωθούν αυτές οι παραβάσεις δεν υπαρχουν ποινικε κυρωσεις η προσπαθεια να διαπιστωθουν αυτες οι ένοπλες δυνάμεις και ομάδες ε, κίνητρα για να σταματήσουν αυτές τις πρακτικές. Επίσης η πείρα αποδεικνύει και τα παιδιά μας το λένε σταθερά ότι μπορούν να γίνουν λιγότερο ευάλωτα μέσω ευρύτερων παρεμβάσεων. Σε πρόσφατες συζητήσεις που είχαμε συναδέλφους στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία με παιδιά που, έχουν να κάνουν, που είχαν ε, στρατολογηθεί από τις ομάδες Εξελέκα και Αντιμπαλάκα κατέστη σαφές ότι όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά δεν ήθελαν να συμμετέχουν. Κάθε παιδί μας έλεγε ότι θέλει να πάει πίσω στο σχολείο και τα μεγαλύτερε ηλικίε θα ήθελαν να μπορέσουν να εργαστούν. Η πρόσβαση λοιπόν στην εκπαίδευση και για τα μεγαλύτερα παιδιά σε δυνατότητα απασχόλησης δεν είναι απλώς μια πρόχειρη λύση. Είναι βασικό σημείο για οποιαδήποτε στρατηγική επανένταξης αλλά και πρόληψης της στρατολόγησης. Όμως ε, πολύ συχνά δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Να συνεχίσω να αναφέρομαι στο παράδειγμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Εκεί εκτιμούμε ότι 6 ε, έως 10.000 παιδιά συμμετέχουν σε ένοπλες ομάδες. Εκεί υπάρχει μόνιμη υποεπένδυση στην ε, εκπαίδευση. Έχει γίνει πολύ πιο έντονο αυτό λόγω των συγκρούσεων. Περίπου δύο τρίτα των σχολείων έχουν κλείσει φέτος. Ορισμένα καταστράφηκαν ή τα έχουν ε, πάρει και τα χρησιμοποιούν οι μαχητές. Η επίσημη οικονομία έχει καταστραφεί. Δύο τρίτα του πληθυσμού ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο τη μέρα. Η ε, καταγραφή στο ληξιαρχείο των γεννήσεων είναι πολύ χαμηλή και τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν τρόπο να αποδείξουν την ηλικία τους. Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έχει υπογράψει, αλλά δεν έχει επικυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο για τη συμμετοχή των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις. Και πατά το, παρά το ότι έχουν γίνει ε, παραπομπές στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνει κάτι στο μέλλον. Η κεντροαφρικανική δημοκρατία μπορεί να είναι ακραία, αλλά δεν είναι καθόλου μοναδική περίπτωση. Παρόμοιες είναι οι συνθήκες σε άλλες ενοπλές συγκρούσει σε κράτη που δεν είναι πολύ σταθερά. Όπω είπαμε, δεν χρηματοδοτείται αρκετά ε, η βοήθεια για τα παιδιά σε ε, επίγουσε συνθήκε. Και σε αυτές τις επίγουσες συνθήκες είναι πιο, τα πιο ευάλωτα τα παιδιά για εκμετάλλευση, στρατολόγηση, σεξουαλική κακομεταχείριση κτλ. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε περισσότερο στα συστήματα προστασία για τα παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σειρά από δυνατότητε για να προστατεύσει τα παιδιά σε συγκρούσει. Αλλά πρέπει ε, όλε αυτέ τι δυνατότητε να εφαρμοστούν με πιο ρωμαλαίο και συστηματικό τρόπο. Η οργάνωσή μα θα ήθελε να τονίσει τέσσερι προτεραιότητε για δράση από το Κοινοβούλιο. Πρώτον, να αυξηθεί η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαπιστώνει και να δράει επί των κινδύνων. Και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καθευτήριες γραμμές για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις και το πρόγραμμα δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αντιπροσωπείες τη Ένωση πρέπει να παρακολουθούν και να κάνουν εκθέσει για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών και να συμμετέχουν σε αυτές τις αποτιμήσεις όχι μόνο ειδικοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και ειδικοί για τα δικαιώματα των παιδιών και για τη βία με βάση το φύλλο. Όλο το προσωπικό στις αντιπροσωπήσεις ιδιαίτερα όταν γίνονται, ε, γίνονται παρεμβάσεις ε, σε ένοπλες συγκρούσεις, να έχουν εκπαιδευτεί όλοι στις ανάγκες των παιδιών. Επίσης, πρέπει να δοθεί περισσότερη προτεραιότητα από πλευράς χρηματοδότησης των μέτρων αυτών. Καλούμε το Κοινοβούλιο να στηρίξει τις προσπάθειες της ε, υπηρεσίας της εξωτερικής δράσης, η προστασία των παιδιών να είναι στο κέντρο των προσπάθειων να καταλάβουμε ότι σώζει ζωές αυτή η παρέμβαση και να δεσμευτούμε ότι θα αυξηθεί χρηματοδότηση για την προστασία των παιδιών σε καταστάσεις επίγουσες και καταστάσεις συγκρούσεων. Τρίτον, σας καλούμε να κάνετε ό,τι μπορείτε για να μην διακόπτεται η εκπαίδευση σε κράτη όπου έχουμε συγκρούσεις να υπάρχει καλύτερη προστασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ιδιαίτερα μετά το ψήφισμά σας του παρελθόντος Μαρτίου για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επαναλάβει τις εκκλήσεις τους στα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν και να εγκρίνουν τις κατευθύνες γραμμές για να προστατεύονται τα σχολεία και πανεπιστήμια κατά, την, ε, κατά τις ένοπλες συγκρούσεις από στρατιωτική χρήση. Έχει, έχουν ολοκληρωθεί αυτέ οι κατευθύνες γραμμέ και θα υποβληθεί στις 16 Δεκεμβρίου στη Γενέβη για να εγκριθεί το 2015. Και κάτι το οποίο νομίζω έχει άμεση σχέση με την εκστρατεία μας, κάτι πολύ συγκεκριμένο που ήδη έχει αναφερθεί. Η Ένωση πρέπει να παίξει καλύτερο ρόλο βοηθώντας τα κράτη να προστατεύουν τα παιδιά μέσω της ε, χρήση προς αυτό το σκοπό της στρατιωτική της βοήθειας. Η προστασία των παιδιών πρέπει να είναι εκπεφρασμένο στόχος της στρατιωτική βοήθειας και η χορήγηση της βοήθειας να εξαρτάται από το κατά πόσο βελτιώνεται η προστασία των παιδιών και κατά την εφαρμογή προγραμμάτων δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Γιύφκα Πέτκοβα που είναι ε, σύμβουλος στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Κυρία Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της κυρίας Μαρινάκη, της Διευθύντριας, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι ευγνώμων για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης σήμερα. Είναι μεγάλη η τιμή να συμμετέχω με τη Λάιλα που συνάντησα στην αρχή της εντολής της, δηλαδή πριν από δυόμιση χρόνια. Αλλά είμαι και περήφανη που μοιράζομαι το έδρανο και με το, τις οργανώσεις Save the Children. Θα ήθελα να σας πω τι ακριβώς κάνουμε σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των παιδιών και ιδιαίτερα των ε, ανήλικων πολεμιστών. Εμείς ε, εφαρμόζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περήφανη που υποστηρίζει αυτή την εκστρατεία της UNICEF. Από την αρχή αυτής της εκστρατείας υποστηρίξαμε τις δραστηριότητες της χώρες σε όλες τις οκτώ χώρες και το στο τσάτα που έχει ε, αφαιρεθεί από τον κατάλογο. Και πρέπει να πω ότι ήμασταν ιδιαίτερα ε, ενεργοί σε αυτό το τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει σκοπό να εντάξει και πάλι τα παιδιά στρατιώτες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ε, στην, ε, στις κοινότητες. Στην εντολή της υπάρχει μια, διαδικασία, μια διαδικασία και συγκεκριμένοι κανόνες. Θα ήθελα να σας παραθέσω ως παράδειγμα την αποστηλή του 2013 όταν ε, θέσαμε ως βασική προτεραιότητα τα παιδιά, τις γυναίκες, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο Επίσης, θέσαμε ως προτεραιότητα την ε, εκπαίδευση πριν από την ανάπτυξη και θα πρέπει να πω ότι υπάρχει και το απαραίτητο υλικό το οποίο είναι κοινό με τις χώρες μέλη και τα Ηνωμένα Έθνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να αυξήσει την προστασία των παιδιών σε, ε, στο επίπεδο της έδρας του και των ε, ενεργειών του. Συνεργαστήκαμε με τη UNICEF, για παράδειγμα, φέτος υιοθετήσαμε ένα πακέτο που αφορούσε τα δικαιώματα των παιδιών. Όχι για να χρησιμοποιηθεί από όλους τους δωρητές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Επιτρέψτε μου επίσης να υπογραμμίσω έναν άλλο τομέα όπου τα ιδιαίτερα και οι συνάδελφοί μας από την Επιτροπή επίσης δραστηριοποιούμε το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην ευημερία. Έχουμε επενδύσει πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ στην πρωτοβουλία Children of Peace, τα παιδιά της ειρήνης, πάνω όπου 108 παιδιά συμπεριλήφθησαν σε αυτό το πρόγραμμα. Αναφερθήκαμε στο Διεθνές ε, Δικαστήριο που και το θέμα της, η καταπολέμηση της ατιμορρησίας για αυτά τα αδικήματα αποτελεί μέρος της δράσης μας. Θεωρούμε ότι το δικαστήριο παίζει καθοριστικό ρόλο και θα ήθελα να, με την ευκαιρία αυτή να σας ενημερώσω ότι ο ρόλος του δικαστηρίου, την εφαρμογή δηλαδή των κατευθυντηρίων γραμμών που αφορούν τα παιδιά στις ένοπλες συγράξεις για υποστήριξη στον ε, ε, εκπρόσωπο υπογραμμίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τις 28 χώρες Βέλη και θεωρήθηκε ένα από τα σημαντικά παραδοτέα το, ε, στην ε, συνάντηση του Λονδίνου. Η Λάιλα αναφέρθηκε στην συνεργασία με περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση οργάνωσε, ε, ασχολήθηκε με μια κοινή διοργάνωση στην Αντισαμπέμπα, όπου ενώσαμε τις δυνάμεις μας με την Παγκόσμια Τράπεζα και την ΟΕΕ βεβαίως. Η πρωτοβουλία αυτή υπήρξε μια ευκαιρία για συζητήσεις σχετικά με την προστασία των παιδιών την, ε, ε, και, τον αφοπλισμό, αλλά και την προστασία των παιδιών σε ε, ε, ε, διαδικασίες, διαδικασίες. Ελπίζουμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας για τη συνεργασία μας και με άλλες οργανώσεις. Εν συντομία θα ήθελα να αναφερθώ στη συζήτηση των, του Συμβουλίου της Ασφαλείας και στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Μετά από αυτή την έκθεση, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριέλαβε και την ε, Νιγηρία στον κατάλογο. Γιατί ε, λόγω της οργάνωσης Μπόκο Χαράμα. Άλλοι τομείς αφορούν τη στρατολόγηση των παιδιών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η UNICEF εφαρμόζουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση χιλίων παιδιών που είχαν σχέση με ένοπλες ομάδες. Επιτρέψτε μου επίσης να υπογραμμίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ε, λύπη της ε, για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν. Την απασχολεί ιδιαίτερα η δολοφονία άμαχων πολιτών στην Συρία και το Ιράκ. Τα παιδιά συνεχίζουν να πλήττονται περισσότερο από κάθε άλλον ε, σαν αποτέλεσμα των συγκρούσεων στη Συρία. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά να τονίσω την πεποίθησή μας ότι το θέμα των παιδιών στις ε, διεθνείς συγκρούσεις θα πρέπει να είναι το βασικό μέλημα των, της διεθνούς κοινότητας, αλλά και δικό μας. Κυρίες και κύριοι, συμπερασματικά, επιτρέψτε μου να σας πω δύο πράγματα. Η Λάιλα ήδη αναφέρθηκε και στην 25η επέτειο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Είναι μια πολύ σημαντική σύμβαση, την οποία, η οποία κυρώθηκε από όλες τις χώρες μέλη και με μεγάλη χαρά θα ήθελα να σας πω ότι θα υιοθετηθούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τα οποία εστιάζονται στις προσπάθειες που έχουν γίνει σε εσωτερικό, ε, ε, ε, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι ο ύπατος εκπρόσωπος ζήτησε από όλες τις αντιπροσωπείες να παρακολουθήσουν την εκστρατή των Ηνωμένων Εθνών 16 μέρες ε, κινητοποίηση. Θα ήθελα να τελειώσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ακούσω με προσοχή τα σχέδιά σας και τα σχόλιά σας σχετικά με τις επόμενες δράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης έχουμε καλέσει έναν εκπρόσωπο από τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν γιατί το Αφγανιστάν είναι μια χώρα που συμμετέχει στην εκστρατεία. Οπότε, αν θέλει, μπορεί να λάβει το λόγο. Sí. Yes. Thank you. Bismillahir Rahmanir uh, Ms. Martinez Ευχαριστώ πολύ στο όνομα του Θεού, του Πολιευσπλάχνου και του Πολιελαίου. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ε, αγαπητοί ε, Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα γιατί εστιάζουμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, τα παιδιά όχι στρατιώτες. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για τη συνδιοργάνωση της σημερινή συνεδρίασης. Ενώ οι παγκόσμιοι ηγέτες δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε κρίσεις πολιτικές, οικονομικές και κρίση ασφαλείας, ε, ξεχνούν να προβλέψουν το μέλλον. Το μέλλον ε, δεν χρειάζεται μόνο προγραμματισμό, σημαίνει ότι πρέπει και να φροντίζουμε όσους θα ζήσουν στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, ε, μία από τις σοβαρές ανησυχίες σήμερα είναι τα παιδιά που χρησιμοποιούνται σε ένοπλες συγκρούσεις σε πολλές χώρες. Στη δική μου χώρα, του Αφγανιστάν, επίσης έχει αναφερθεί μεταξύ των χωρών αυτών. Ε, πριν όμως ε, ασχοληθώ με το θέμα αυτό στο Αφγανιστάν, θα ήθελα να αναγνωρίσω και να εκτιμήσω ε, την προσφορά της κυρίας Λέιλα Ζερούγκη και την προσφορά, την προσφορά της ειδικότερα στο θέμα των παιδιών και της προστασίας αυτών από τις ένοπλες συγκρούσεις, τη UNICEF και τη Σώστε τα παιδιά ώστε να απαρεμποδιστεί ε, και να εξαλειφθεί πλήρως η στρατολόγηση των παιδιών μέχρι το 2016. Η εκστρατεία ήταν πάρα πολύ επιτυχής και αποτελεσματική στο Αφγανιστάν. Εξοχότητες. Το άρθρο 54 του Συντάγματος του Αφγανιστάν αναφέρει την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών. Το άρθρο 49 αναφέρει ρητός ότι η εξαναγκαστική εργασία απαγορεύεται, η εξαναγκαστική εργασία των παιδιών. Ε, αυτά τα άρθρα είναι η βάση της δέσμευσή μας ε, για, ε, τη για την συνεργασία μας με τον ΟΗΕ στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας. Είναι πάρα πολύ επαγγελματικές οι δικές μας εθνικές στρατιωτικές δυνάμεις. Δεν στρατολογούν παιδιά. Παρόλα αυτά δεν αρνούμε το γεγονός ότι υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν στρατολογηθεί παιδιά από την τοπική αστυνομία και είναι 14 τα παιδιά που έχουν αναφερθεί ε, σε έκθεση του ε, Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Συμβούλιο, της, ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα ήθελα να αναφερθώ λοιπόν στην έκθεση 339 στην οποία αναφέρεται ότι σε μια περίπτωση, σε μια επαρχία λαχμών ε, συνελήφθησαν 21 παιδιά από ηλικίας από 7 ετών ε, στην, όταν πήγαιναν στο Πακιστάν για επίθεση αυτοκτονίας ε, και εκπαίδευση από τους Ταλιμπάν. Αυτά τα παιδιά είχαν μια καλή, δεν γνώριζαν τι θα τους συμβεί ε, όταν, πήγαιναν, όταν θα πήγαιναν στο Πακιστάν. Ε, οι Ταλιμπάν έχουν στρατολογήσει πολλά παιδιά, εκατοντάδες και από το Αφγανιστάν και από το Πακιστάν. Τους έκαναν πλήση εγκεφάλου και τα χρησιμοποιούσαν ε, κατά των αφγανικών ε, δυνάμεων ασφαλείας. Ε, μερικές φορές ε, παιδιά που παίρνουν από τους μαντρασάδες χρησιμοποιούνται ως βομβιστές αυτοκτονίας. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς στρατολογούνται τα παιδιά αυτά. Ε, μπορεί να στρατολογηθούν τώρα και να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική ένοπλη σύγκρουση. Ένας από τους κύριους λόγους είναι η έλλειψη πρόσβασης εκπαίδευσης. Οι τρομοκρατικέ οργανώσεις ε, συχνά ε, καίνε σχολεία σε πολύ μακρινές περιοχές και μετά προ, προ, προτείνουν θρησκευτική εκπαίδευση στι θρησκευτικέ οικογένειες, ε, στα, ε, θρησκευτικά, θρησκευτική εκπαίδευση στι οικογένειες, ε, οι οποίες δεν μπορούν να θρέψουν και να ντύσουν τα παιδιά τους. παίρνουν λοιπόν τα παιδιά και τους λένε ότι θα τα πάνε σε οικοτροφία, τα οποία θα, στα οποία θα ντύσουν και θα θρέψουν τα παιδιά τους ότι θα τους δώσει τη δυνατότητα εκπαίδευσης ε, καλύτερης ε, και πρόσβαση στην εκπαίδευση που η κυβέρνηση είναι ανίκανη να τους παρέχει. Σε σχέση τώρα για, σε σχέση με τη σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών του ΟΗΕ, είναι ισχυρή και θετική η δέσμευση του Αφγανιστάν. Έχει σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με τη συμμόρφωση ε, προς το σχέδιο δράσης για να λήξει ε, και για να υπάρξει καταπολέμηση της στρατολόγησης παιδιών. Η κυβέρνηση του Αφγανιστάν θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης σύμφωνα με τον οδικό χάρτη 15 σημείων ε, του Αυγούστου του 2013. Το Αφγανιστάν έχει υποβάλει την τρίτη έκθεσή του το Μάρτιο του 2014 ε, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα λεπτομερή βήματα προς την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Και θα ήθελα επίσης να πω ορισμένα πράγματα για την ε, ε, ε, επίσκεψη του Προέδρου του Αφγανιστάν στο Ευρωπαϊκό, στις Βρυξέλλες και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιν Σούλτς και μίλησε για αμοιβαίο ενδιαφέροντος θέματα μαζί του, ειδικότερα για τα δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών, ένα θέμα που ήταν πολύ υψηλά στις προτεραιότητες της συζήτησής τους. Τα παιδιά είναι η ίδια η ζωή. Πρέπει να είμαστε ε, καλά, καλοί μαζί τους, πρέπει να, τους, να τα βοηθήσουμε να ε, νιώθουν ασφαλή μέχρι το τέλος της ζωής τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μήπως συνάδελφοι θέλουν το λόγο? Α, ποιος? Παρακαλώ. Δεν με σπάκε. έγιος πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, πριν από λίγο ακούσαμε ορισμένα ομολογουμένως εντυπωσιακά, ενδιαφέροντα και σαφώς εξοργιστικά πράγματα από διακεκριμένες ομιλήτριες και διακεκριμένους ομιλητές που έχουν σχέση με τη χρησιμοποίηση των παιδιών ως στρατιωτών σε πολεμικές συγκρούσεις για τη βία που ασκείται πάνω σε αυτά για τις ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, για τις επιπτώσεις που θα έχουν στην ψυχική τους κυρίως υγεία η χρησιμοποίησή τους σε πολεμικές συγκρούσεις και πολλά και διάφορα. Και ερωτώ με, ποια είναι η θέση που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ο ΙΕ απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Ευχολόγια, υψηλού επίπεδου φιλοσοφικές αναλύσεις συζητήσεις επί συζητήσεων με τις κυβερνήσεις των κρατών που παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών, τα χρησιμοποιούν σε πολεμικές συγκρούσεις και δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε τις νοθεσίες αλλά ούτε ενδεχομένως και τις αυστηρές προειδοποίησεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γιατί άραγε αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα με τόσο μεγάλη υποκρισία. Γιατί δεν λαμβάνουμε αυστηρά μέτρα εναντίον όλων αυτών που παραβιάζουν με αυτόν τον τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχετε ακούσει να επιβληθούν οικονομικά ή άλλης φύσεως μέτρα εναντίον των κυβερνήσεων αυτών που χρησιμοποιούν τα παιδιά σε πολεμικές συγκρούσεις. Έχετε ακούσει να κληθούν οι πρόεδροι των κυβερνήσεων αυτών στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή στο Δικαστήριο Εγκληματιών Πολέμου για να απολογηθούν ως κατηγορούμενοι. Δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Πολλές φορές εξαντλούμε την αυστηρότητά μας για να αντιμετωπίσουμε πολιτικούς μας αντιπάλους επειδή αυτά τα οποία λένε είτε δεν μας αρέσουν είτε τα θεωρούμε επικίνδυνα και αδιαφορούμε για πραγματικά επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες προσβάλλουν και τις αρχές της δημοκρατίας και παραβιάζουν και τις αρχές του ανθρωπισμού. Βλέπετε, ευτυχώς ή δυστυχώς, τα παιδιά δεν ψηφίζουν ούτως ώστε να προσδοκούμε σε κάποιο άμεσο πολιτικό όφελος. Και εκείνο το οποίο πραγματικά κάνουμε είναι να σκουπίζουμε και να βάζουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί πιστεύοντας ότι έχουμε επιτελέσει το καθήκον μας. Και η ζωή συνεχίζεται δυστυχώς ως εφιάλτης για αυτές τις ανθρώπινες υπάρξεις που δεν φαίνεσαι τίποτε για εκείνο το οποίο υφίσταται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ τους ομιλητές μας για όλες τις λεπτομέρειες που μας έδωσαν σήμερα. Μας παρουσίασαν αυτό το τόσο σοβαρό φαινόμενο, τη χρήση παιδιών ως στρατιωτών. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Χθε το βράδυ, κατά σύμπτωση, είδα ένα ντοκιμαντέρ στην φλαμανδική τηλεόραση για τα προγράμματα αποκατάσταση και επανένταξη των παιδιών αυτών στην Ουγγάντα. Και οι ιστορίε, οι εικόνε που είδα ήταν πραγματικά τρομακτικέ. Η κυρία Τίμερμαν έχει εργαστεί ε, εδώ και χρόνια για τέτοια προγράμματα στην Ουγκάντα. Θα είχα λοιπόν μερικές ερωτήσεις και μερικές σκέψεις. Υπάρχει πολύ καλή διάθεση και πολλές πρωτοβουλίες. Αλλά παρά όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, τι διαπιστώνουμε και στη χώρα μας και σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Διαπιστώνουμε ότι πολλοί γίνονται όλο και πιο ακραίοι και πάνε στο Ιράκ και τη Συρία για να πολεμήσουν. Για να πολεμήσουν ως μέλη του Ισλαμικού κράτους, του IS και παίρνουν και παιδιά μαζί τους. Τα οποία μετά τα βλέπουμε στο βίντεο. Σε βίντεο, συγγνώμη, στο ίντερνετ όπου κουνάνε ανθρώπινα κεφάλια ως τρόπεα. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει, αλλά είναι πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καινούριο φαινόμενο που αφορά πολύ πιο άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον θα έπρεπε να το συζητάει. Θα πρέπει η αντίδρασή μας να είναι η αρμόζουσα προς αυτό το καινούριο φαινόμενο που θεωρώ ότι είναι ένα κοινωνικό πλέον φαινόμενο. Βεβαίω θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ε, σχολείων, των εκπαιδευτικών. Επίσης ε, περισσότερο κοινωνικό έλεγχο θα χρειάζεται. Επίση περισσότερε ε, δυνατότητε, οικονομικέ και κοινωνικέ σε αυτού που δεν αισθάνονται σαν να είναι στο σπίτι τους ε, για οποιοδήποτε λόγο στις χώρες μας. Δεν άκουσαν να μας λένε τίποτα οι ε, ειδικοί. Επίσης, ε, ξέρω ότι υπάρχουν πολλές διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Βεβαίως, υπάρχουν. Αλλά αρκούν για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Δεν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ορισμένες από αυτές τις συνθήκες στην ουσία έχουν περιπέσει σε αχρησία. Θα έπρεπε να ανανεωθούν, να εξυγχρονιστούν. Τι μπορεί να κάνει η Ένωση για αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, η Σύμβαση της Γενέβης, όπου αναφέρονται μια σειρά από για να καθορίσουν τι σημαίνει ε, μαχητής έναντι του αμάχου πληθυσμού. Όμως ε, Κανένα από αυτά τα κριτήρια, αν διάβασα καλά, δεν αναφέρεται στην ηλικία του μαχητή. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να εξυγχρονιστεί η σύμβαση. Και γενικότερα και άλλε συμβάσει. Δεν θα έπρεπε όλε αυτέ να εξυγχρονιστούν, να προσαρμόσουν. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Και τέλο. Βλέπω εδώ το κατάλογο των χωρών όπου υπάρχει αυτό το τρομερό πρόβλημα, αυτή η μάστιγα. Και τι διαπιστώνω. Ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο σημαντικό στα αποτυχημένα κράτη, τα κράτη που έχουν καταρρεύσει. Στα κράτη αυτά η φτώχεια είναι ακραία, υπάρχουν ένοπλες ε, σειράξεις, που είναι φυσικά η ρίζα του φαινομένου. Ε, ο κατάλογος έχει χώρες ε, διαφορετικού χαρακτήρα. Ορισμένα κράτη που ήταν προηγουμένως στο κατάλογο ευτυχώς έχουν απαλληφθεί, αλλά προστίθεται δυστυχώς νέα. Και νομίζω ότι η κυρία Withers το είπε είπε ότι πρέπει να δούμε σε ποιες είναι οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος. Ότι είναι ζωτικό αυτό. Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε περισσότερα από αυτού. Βεβαίως. Εύκολα μπορούμε να δούμε κάποιες περιφέρειες όπου μπορούμε να προβλέψουμε με μεγάλη πιθανότητα ότι θα πέσουμε μέσα, ότι θα προκύψουν συγκρούσει. Αλλά τι θα κάνουμε μετά, ούτω ώστε η κατάσταση να μην επιδεινωθεί και να μην προκύψει λοιπόν το πρόβλημα. Το πρόβλημα τη στρατολόγηση παιδιών. Καλή είναι η πρόβλεψη, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε μετά για να αποφύγουμε οι προβλέψει μα να επαληθευθούν. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε το χειρότερο δηλαδή. Τι μπορούμε να κάνουμε ως πρόληψη των ενόπλων συγκρούσεων. Ευχαριστώ άλλη μια φορά για τις παρουσιάσεις σας και για τις απαντήσεις που θα μου δώσετε. Ευχαριστώ λέει και πρόεδρος κύριε Μάκερ. Ο κύριος Άουστρεβίτσιους. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το πάνελ που μας βοήθησε να καταλάβουμε το πώς ακριβώ έχουν τα πράγματα με τα παιδιά που εμπλέκονται σε ματηρούς πολέμους. Όσοι στρατολογούν και οργανώνουν την ένταξη παιδιών στρατιωτών διαπράττουν ένα σοβαρό έγκλημα. Θα μπορούσε κάποιος από εσά να πει το εξής. Εκλήθη κάποιος ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης με την κατηγορία της διάπραξης ενός εγκλήματος. Ποια είναι η γενικότερη πρακτική του Διεθνούς Δικαστηρίου σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Μπράντα. Συγγνώμη. Συγγνώμη πρώτα στον κύριο Χολή. Μετά η κυρία Μπραντ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντεμισμέκερ, έχετε δίκιο. Ο πόλεμος των παιδιών άρχισε στην Ευρώπη και εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε δεσμευθεί πολύ. Περίπου 1% 8 ευρωβουλευτές ε, σήμερα ε, έχει δεσμευθεί. αλλά έχει ξεκινήσει υπάρχει και στην Ευρώπη. Και το δράμα που βλέπουμε ε, είναι, αρχίζουν ε, οι, οι κραυγές απελπισίας. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, όπως είπατε κι εσείς, ε, ποιο, τι, πρόληψη μπορούμε να έχουμε στις χώρες στις οποίες εσείς μέσω των αντιπροσωπιών σας έχετε την επιρροή. Και πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά πρωταθλήτρια. Η κυρία Μογκερίνη την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια, κατόπιν ψηφίσματος των Ευρωβουλευτών, δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί μέσω τη εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα των παιδιών. Και είναι μοναδικό αυτό το φαινόμενο στον κόσμο. Κατόπιν λοιπόν του δικού σα. Ε, ε, ψηφίσματος ε, είπε ότι ε, πρέπει οπωσδήποτε να επικυρωθεί αυτή η σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο θα είναι πολύτιμο όλες αυτές οι πτυχές της υφόρου ε, ανάπτυξης, ε, της καταπολέμησης της ε, ανεργίας είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει να συνδεθούν με αυτό το θέμα. Μία χώρα που αναπτύσσεται χωρίς να επενδύει, να επενδύει στα παιδιά είναι μία χώρα που δεν επενδύει, δεν, δεν αναπτύσσεται. τώρα, για το πολιτικό επίπεδο. Έχει στο διεθνές προσκήνιο επιρροή και ε, κάποια βαρύτητα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προχωρήσει το θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο και της ε, συγκεκριμένης εκστρατείας παιδιά όχι στρατιώτες ε, μέσω των διαφόρων μέσων και του ΟΗΕ αλλά και μέσω άλλων οδών είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Ε, η κατάσταση είναι και πολιτικής φύσεως. Οι συνάδελφοι από το Αφγανιστάν το γνωρίζουν. Στο Τσάντ, στο Κονγκό είναι καταρχάς πολιτικό το θέμα. Χρειάζεται μια δέσμευση και για να υπάρξει αυτή η δέσμευση, χρειάζεται κινητοποίηση δικτύων και πολλές πολιτικές δυνάμεις που θα συνεργαστούν. Και γι' αυτό ε, υπάρχει ανάγκη ε, δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε σήμερα να δούμε μέσω των κοινωνικών δικτύων να επιτρέψουμε στραφολόγηση ακόμα πιο αποτελεσματική. Ε, να μην σας πω ότι έγιναν και πάρα πολλές μέλη στα διαφημιστικές εκστρατείες ε, από συγκεκριμένες τρομοκρατικές ομάδες. Πρέπει να είμαστε ε, πολυάριθμοι, πιο πολυάριθμοι από ότι είμαστε σήμερα στη συγκεκριμένη αύξηση, γιατί έχει αρχίσει αυτός ο πόλεμος και είναι μια, ένας πόλεμος που δεν είναι καθόλου συμβατικός. Θα γίνει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα γίνει μέσω της πολιτικής επιρροής ε, μέσω δικτύων που έχουν ε, εδώ και πολλά χρόνια αναπτυχθεί ε, δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή αυτή η νέα μορφή βίας. Γι' αυτό σας ζητούμε ε, σε εσά, ε, ευρωβουλευτέ, να μην δείξετε καμία ανοχή. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να τύχει καμία ανοχή. Αυτό είναι το μήνυμά μας και νομίζουμε ότι είναι ένα καταρχάς πολιτικό μήνυμα, ένα μήνυμα συνεργασία σε όλα τα επίπεδα κυβέρνηση, κοινωνία των πολιτών, ε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των κοινοβουλίων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βίδες από τη σώστα τα παιδιά. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ή δύο σημεία σχετικά με την παρέμβαση αυτή και Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει ένα διαθέσιμο πακέτο έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση σε ό,τι αφορά αυτά που έχουν αποφασιστεί. Το πακέτο αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ξεκινάει με θέματα που αφορούν την επικοινωνία, περνάει στις κληρώσεις και νομίζω ότι συμβάλλει στον, για να μπορέσει να υπάρξει αξιοπιστία θα πρέπει να υπάρξει μία παρακολούθηση για να δούμε αν υπάρχει εφαρμογή. Το 2012 ψηφίστηκε ε, ένας ε, νόμος και μετά υπήρξε ένα πρόγραμμα δράσης για, την, ε, για τους ανηλίκους μαχητές. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν όλα αυτά. Ετέθη το ερώτημα σχετικά με το αν αρκούν οι υπάρχουσε συμφωνίες. Η απάντηση για μένα είναι και ναι και όχι. Το κανονιστικό πλαίσιο είναι επαρκές. καθώς και το πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε άλλους τομείς όμως θα πρέπει να δούμε κατά πόσον η προστασία που παρέχει το υπάρχον πλαίσιο είναι επαρκής. Αναφέρθηκα συγκεκριμένα στην στρατιωτική χρήση των σχολείων. Είναι κάτι που αποθαρρύνεται αλλά δεν απαγορεύεται από το ανθρωπιστικό δίκαιο. Το θέμα είναι ότι η χρήση των σχολείων από στρατιωτικέ ομάδες τα καθιστά ευάλωτα σε επιθέσεις και αυτό έχει μια άμεση επίπτωση στην ασφάλεια των παιδιών. Αλλά επηρεάζει και την δυνατότητα ε, που έχουν να μορφωθούν. πω ότι θα πρέπει να υπάρξουν κατευθυντήριοι γραμμές για τη στρατιωτική χρήση των σχολείων. Θα υποβληθούν και θα, είναι, θα τεθούν προς έγκριση αργότερα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να δείξω και αφορά τη χρήση εκρηκτικών όπλων. Αυτά είναι συμβατικά όπλα. Το πρόβλημα όμως με αυτά τα όπλα είναι ότι όταν χρησιμοποιούνται σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές, η πλειοψηφία των θυμάτων προέρχονται από τον άμαχο πληθυσμό και ιδιαίτερα από τα παιδιά. Εμείς δεν αναζητάμε την κατάργησή τους, θα πρέπει όμως να μας απασχολήσει το κατά πόσον η χρήση τους θα μπορούσε να περιοριστεί σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις. Ετέθηκε το θέμα του πώς πρακτικά αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους. Υπάρχουν πολλά ε, πολλές πρακτικές ε, δράσεις που θα μπορούσαν να αναλυθούν. Το νομικό πλαίσιο δεν είναι μια πανάκια. Είναι σημαντικό όμως το να υπάρχει γιατί δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο είναι δυνατόν να δοθεί προστασία. Αυτό το επίσης είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει ένα έγγραφο που να αποδεικνύει την ηλικία των παιδιών. Πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν κάποιο πιστοποιητικό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί η ηλικία των παιδιών. Ετέθησαν θέματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη, την εκπαίδευση. Όλα αυτά τα θέματα είναι καθοριστική σημασία. Όπως είπα στην παρουσίασή μου, πολύ συχνά τα παιδιά αυτά δεν έχουν εναλλακτικέ λύσεις, δεν έχουν επιλογές, δεν υπάρχει εναλλακτικό δρόμος. Αναζητάνε κάτι άλλο. Δεν θέλουν να ενταχθούν σε αυτές τις ομάδες, αλλά δεν τους παρέχεται κάποια εναλλακτική λύση. Υπάρχει και ένας άλλος τομέας ε, που θα ήθελα να εξετάσουμε που αφορά το γιατί στρατολογούνται τα παιδιά. Πέρα από το γιατί θα πρέπει να δούμε το πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν τυπικές διαδικασίες στρατολόγησης. Υπάρχει κάποιος έλεγχος αυτών των διαδικασιών. Υπάρχει κάποια ποινικοποίηση των παράνομων τρόπων στρατολόγησης, κάποια παρακολούθηση. Υπάρχουν πολλές πρακτικές δράσεις που θα μπορούσαν να αναλυθούν, αλλά δεν υπάρχει ε, τρόπος για να τα αντιμετωπίσουμε ε, εκ των ενόντων. Ευχαριστώ κυρία Σερούγη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που επιδείξατε. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας, θέλω να τονίσω. Και εμένα, και εμένα μου συμβαίνει ορισμένες φορές αγανακτό, εξοργίζομαι, γιατί πραγματικά λέει κανείς πώς είναι δυνατόν να συνεχίζονται αυτά τα πράγματα. Αλλά θα ήθελα να είμαι θετική σήμερα, να έχω θετική, δεν θέλω να σας ε, απογοητεύσω σήμερα, να σας στενοχωρήσω. Αν δούμε στον κατάλογο ότι μόνο 7 χώρες αναφέρονται για τη στρατολόγηση παιδιών, είναι ήδη κατόρθωμα. Όπως ξέρετε υπάρχουν 194 κράτη στον πλανήτη μας. Και ένα από αυτά, το Αφγανιστάν, εκεί είδαμε ότι δεν αναφέρεται ο στρατός, αλλά μια τοπική αστυνομία. Άρα το θέμα είναι να μπορούμε να είμαστε παρόντες ε, επιτόπου στα χωριά και συνεργαζόμεθα στενά για να μην συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει συνένεση. Δεν υπάρχει ούτε ένα κράτο που να λέει δεν είναι δικό σα θέμα, εγώ στρατολογώ παιδιά. Πριν το κάνανε, τώρα δεν το κάνουν. Έγινε λοιπόν μια δουλειά από αυτού. Τώρα, ξέρετε, από τι 59 οργανώσει ε, που στρατολογούν παιδιά, 51 είναι ένοπλε ομάδε. Ορισμένοι δεν θέλουν ούτε καν να μα ακούσουν, Όπω είδαμε στην ταινία που δείξαμε, στο βίντεο. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε μέτρα εναντίον των ομάδων αυτών. Πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη όπου υπάρχει πολιτική βούληση, ούτω ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα ατιμορρησίας. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά μπορεί να κάνει. Πολύ συχνά είδαμε ότι τα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν αυτά τα προβλήματα είναι σε δύσκολη θέση. Δεν υπάρχουν θεσμοί. Είναι υποχρεωμένα τα κράτη αυτά να διαπραγματεύονται με ένοπλες ομάδες που απαιτούν να γίνουν τμήμα των ενόπλων δυνάμεων. Ε, εγώ ήμουν στο Κονγκό όταν μια ένοπλη ομάδα που είχε τρομερά μεγάλο αριθμό παιδιών στρατιωτών έγινε τμήμα των ενόπλων δυνάμεων. Και δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να γίνει ένας έλεγχος για να ε, απολυθούν αυτά τα παιδιά. Και τώρα, μετά από τέσσερα χρόνια, το Κονγκό λέει δεν θα δεχθώ άλλα παιδιά, δεν θα δοθεί αμνηστία και θα διωχθούν αυτοί που στρατολόγησαν παιδιά. Αυτή η δέσμευση πρέπει να, βεβαιώσουμε, να βεβαιωθούμε ότι θα εφαρμοστεί. Γιατί ορισμένε φορέ η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ορισμένε δυσκολίε και κάνει υποχωρήσει. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε, τόσο ώστε η δέσμευση, η δέσμευση που αναλήφθηκε θα εφαρμοστεί ακόμη και αν ε, κάποιες ένοπλες δυνάμεις ε, ενταχθούν, κάποιες ένοπλες ομάδες ενταχθούν σε ένοπλες δυνάμεις του κράτους να μην ενταχθούν ατιμωρητοί αυτοί που στρατολόγησαν παιδιά. Εκεί που υπάρχει η πολιτική βούληση πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αλλά εκεί που δεν υπάρχει, όταν κάποιοι δεν θέλουν να λάβουν μέτρα, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εμείς άλλες δυνατότητες. Τότε πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε. Επίσης, ε, τέθηκε ένα ερώτημα. Τι μπορεί να κάνουμε για αυτήν την ριζοσπαστικοποίηση των νέων και των παιδιών. Βλέπουμε τις εικόνες από το Ισλαμικό κράτος ε, μέσω των κοινωνικών μέσων. Αλλά και στο Κονγκό. Και εκεί που έχουμε το στρατό του Κυρίου Επίση στρατολογούσαν παιδιά, δεν χρησιμοποιούσαν κοινωνικά μέσα, αλλά υποχρέωναν τα παιδιά να σκοτώσουν, να βιάσουν κτλ. Και τον Μποκοχαράμ το κάνει. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι όπου υπάρχουν ομάδε που στρατολογούν παιδιά, τα παιδιά υφίστανται αυτά που μας δείχνει το Ισλαμικό κράτος και ακόμη πιο πολλά. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Πρέπει να απαντήσουμε με ευφυή τρόπο να μην δώσουμε λάθος απαντήσεις. Γιατί η απάντηση πρέπει να σημαίνει την εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων και να μην στιγματίζονται τα παιδιά αυτά. Στόχος μας πρέπει να είναι αυτό που λέω να αποξηρανθεί ο βάλτος. Έτσι το αποκαλώ. Δηλαδή πρέπει να αφαιρέσουμε το υπόστρωμα που επιτρέπει να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Πρέπει να κάνουμε μια εργασία ευαισθητοποίησης, επανένταξης, μια εργασία ανάπτυξης. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να σκεφτούμε και σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περιοχή να δούμε τι είναι το πιο κατάλληλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εργαστεί και ως Ένωση και επίσης και άλλα κράτη μπορούν να βοηθήσουν. Εγώ είμαι Αλγερινή Ξέρω ότι και στην ε, περιφέρειά μου υπάρχουν νέοι που πάνε, που στρατολογούνται. Και εκεί προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στη χώρα μας για να μην συνεχίζεται αυτό το φαινόμενο. Πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε κάθε νομιμοποίηση από τα κράτη αυτά. Να τους πούμε όχι, δεν εκπροσωπείτε το Ισλάμ, δεν εκπροσωπείτε την κοινότητά μου. Είστε εγκληματίες. Αυτό είναι σημαντικό. Αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε σημειώσει πρόοδο. Επίσης ε, Τέθηκε το ερώτημα, δεν είναι παρόν νομίζω εκείνος που το έθεσε, αν υπάρχουν παραδείγματα αποφάσεων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη στρατολόγηση παιδιών. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ήταν η πρώτη απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ήταν η υπόθεση Λουμπάγκα που μόλις επικυρώθηκε από το εφετείο. Για τη στρατολόγηση παιδιών ήταν. Ο Τσάλς Τέιλορ, πρώην πρόεδρος της Λιβερίας, καταδικάστηκε για στρατολόγηση παιδιών. Ο Τόμας Μποσκονταγκάντα επίσης ε, έχει, του έχει απαγγελθεί κατηγορία ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ε, και ο Ζερμέν Κατέγκα. Όλα αυτά τα άτομα μπόρεσε το δικαστήριο να τους απαγγείλει κατηγορία με βάση την ευθύνη του διοικητή. Είπε το δικαστήριο, εφόσον στην μονάδα την οποία διοικείται υπάρχουν παιδιά, έχουν παιδιά και δεν έχουν απολυθεί, είστε υπεύθυνο. Με βάση αυτή την αρχή το δικαστήριο του απήγγειλε κατηγορίε. Αυτό είναι καλό βέβαια. Αλλά καλύτερα θα ήταν τα εθνικά δικαστήρια να το έχουν κάνει. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν διαπιστώνω, για παράδειγμα, στην έκθεση που μόλι έλαβα από το Υπουργείο Άμυνα του Κονγκό, Χαίρομαι πολύ όταν βλέπω ότι ο επικεφαλή της τάδε ομάδας, ο αρχηγός Ντενιατούρα, ο αρχηγός Μάι Τσιτάνη, όλοι αυτοί ε, κατηγορούνται για, δηλαδή του έχει απαγγελθεί κατηγορία για στρατολόγηση παιδιών. Αυτό έχει γίνει. Τώρα δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά δεν θέλω να αποφύγω τι ερωτήσει. Τώρα, τέθηκε μία ερώτηση για το νομικό πλαίσιο, το διεθνέ νομικό πλαίσιο. Αν επαρκούν οι συμβάσει και συνθήκε έχουμε επαρκεί δυνατότητε μέσω αυτών. Εγώ δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη. Γιατί η ελάχιστη ηλικία κάτω από την οποία ε, είναι παράνομη στρατολόγηση είναι 15. Θα προτιμούσα 18. Χαίρομαι πολύ που η Αφρικανική Χάρτα για την Ευημερία των Παιδιών αναφέρει 18. Πολλές χώρες του Νότου ορίζουν 18 ενώ στο βορρά η ελάχιστη ηλικία ορίζεται 16, στα 16-17. Θα μπορούσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι θέτουμε ως απόλυτο όριο το 18, τα 18. Αυτό θα ήταν πολύ καλό. Διότι η στρατολόγηση παιδιών είναι διεθνές έγκλημα, αν είναι κάτω από 15. Και δεν έχουμε πιο αυστηρή νομοθεσία ε, επειδή ορισμένε μεγάλε χώρε ήθελαν να συνεχίσουν να μπορούν να στρατολογούν παιδιά 16 ετών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζερούγκη. Και τώρα, για να κλείσει την ε, συνάντηση, θα δώσω το λόγο στον κύριο Πλένκοβιτ. Ευχαριστώ πολύ. Στα κροατικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τους προσκεκτικούς για αυτό το σημαντικό θέμα σε σχέση με την εκστρατεία παιδιά όχι στρατιώτες. Είναι πραγματικά ένα θέμα παγκοσμίου σημασίας. Ε, γι' αυτό ακριβώς υποστηρίξαμε την πρωτοβουλία της κυρίας Βαλεντιάνο για να συζητηθεί το θέμα αυτό ενώπιον της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την εκστρατεία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες να εξασφαλίσουμε ότι η εστίαση γίνεται σε αυτό το σοβαρό θέμα της στρατολόγησης παιδιών ε, στις ένοπλες συγκρούσεις. Δείχνει λοιπόν όλη η συζήτηση ότι υπάρχουν κάποιες χώρες σε αυτό τον κόσμο που δεν λειτουργούν καλά που είναι πολύ αδύναμες που δεν έχουν αρκετά ισχυρούς θυσμούς προ, ώστε να αποφευχθούν ε, τέτοιου είδους πρακτικές και την κακοποίηση των παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις. Γι' αυτό ακριβώς η εκστρατεία αυτή, όπως και στοχευμένες δραστηριότητες του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ σημαντικές είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής μας και πρέπει να αποτελέσει ε, σημείο εστίασης συνεχούς, γιατί είναι κάτι που έχει να κάνει με τις θεμελιώδεις αξίες που υπερασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλές συμφωνίες ε, οικονομικής ενίσχυσης και άλλες ε, μορφές ενίσχυσης και πιστεύω ότι αυτό το θέμα πρέπει πάντοτε να εξετάσετε στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, γιατί το τελικό αποτέλεσμα αυτών των συμφωνιών πρέπει να είναι αποτέλεσμα της τάσης που έχει η άλλη πλευρά για το θέμα της στρατολόγησης των παιδιών. Πρέπει λοιπόν να είναι πολύ στοχευμένη η αντιμετώπιση του προβλήματος. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η άποψη της εξωτερικής υπηρεσίας ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, το θέμα της συνεργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θεωρηθεί παγκόσμιο αυτό το θέμα. Πρέπει να είναι δυναμική και συνεχής η συζήτηση στο πλαίσιο όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός αυτής. Θα ήθελα μία ακόμη φορά λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες εκ μέρους του κυρίου Μπροκ. Μία ακόμη φορά να επαναλάβω ότι υποστηρίζω απολύτως την εκστρατεία ε, «Παιδιά όχι στρατιώτες» και τις προσπάθειες ε, της κυρίας Ζερούγκη αλλά και των υπολείπων προσκεκλημένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, λίγη η ακρόαση.